μέτρα της Επιτροπής προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση στην υπόθεση ΤΑΦ 521 14 Σουηδία κατά Επιτροπής. Υποχρέωση θέσπισης κριτηρίων για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, παρεμβαλλόμενες ουσίες. Προφορική ερώτηση. Αυτό είναι το επόμενο θέμα. Ο λόγος. Καταρχήν στους συντάκτες. Την κυρία Γκούτελαντ. Δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Οι διαταράκτες ε, απαντώνται παντού στην καθημερινή ζωή. Στα τρόφιμα, τις σκευασίες, τα παιχνίδια των παιδιών, στο πόσιμο νερό. Συνδέονται μάλιστα, βάσει ερευνών, με σειρά ασθενών όπως ο διαβήτης, ο καρκίνος και με αυξημένους κινδύνους για τη γονιμότητα πρόκειται για μια πολύ ανισχυτική κατάσταση. Παιδιά, μωρά, έμβρια εκτίθενται σε αυτές τις ουσίες τα αποτελέσματα των οποίων εμφανίζονται μόνο αργότερα στη ζωή. Ανησυχούμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τους νομοθέτες να δεσπίσουν σχετική νομοθεσία. Οι σοσιαλιστές είναι στην πρωτοπορία αυτών των ετούντων. Υποχρεώσαμε και είμαστε περήφανοι γι' αυτό την Κομισιόν να τηρήσει τις υποχρεώσεις της. Διότι αυτή έχει την υποχρέωση να, θέσει, να θεσπίσει επιστημονικά κριτήρια για τις ουσίες αυτές. Όμως, η Κομισιόν καθυστερεί να θέσει σε ισχύ τη σχετική νομοθεσία. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από την σχετική απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου. Χρειάζεται λοιπόν να θεσπιστούν επιστημονικά κριτήρια. Εν απόσία αυτών και μη νομοθετώντα, νομοθετώντας, η Κομισιόν παραβιάζει την ενωσιακή νομοθεσία και αυτό είναι παράδεκτο. Η Κομισιόν μας λέει τώρα ότι θα λάβει μέτρα προσπαθώντας να θεραπεύσει την έλλειψη νομοθεσίας. Ελπίζω ότι θα σταματήσει να καθυστερεί, να κολλησιεργεί η Κομισιόν σχετικά με, την, τους κανόνες για τους ενδοκρινικούς διδαράκτες. Κομισιόν, αναλάβατε την ευθύνη σας ενώπιον των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει των συνθήκων, αυτή είναι η πρώτη ευθύνη σας. Ελπίζω αυτή τη φορά να έχουμε μια σαφή απάντηση από την Κομισιόν. Πρόεδρος, επόμενος ο ο κύριος Χελμπράντη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν ζητούσετε από κάποιον να ιεραρχήσει τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή του, το πιο πιθανό είναι ότι η υγεία θα ήταν στην κορυφή αυτού του καταλόγου. Και αυτό είναι το αντικείμενο μας σήμερα. Η υγεία. Γιατί ακριβώς η υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Το θέμα που έχουμε εδώ μπροστά μας είναι σαφέστατο. Έχουμε έναν κανονισμό, έναν, ένα νομικό κείμενο και σε αυτό το νομικό κείμενο υπάρχει μια συγκεκριμένη υποχρέωση για την Κομισιόν να θεσπίσει επιστημονικά κριτήρια ω τον Δεκέμβριο του 2013 για του ενδοκρινικού διαταράκτε. Δεν είναι γραμμένο στα κινέζικα, είναι γραμμένο σε όλε τι ε, επίσημε γλώσσε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκύπτει λοιπόν σαφώ η προθεσμία. Δεκέμβριο του 2013 η Κομισιόν έπρεπε να είχε θεσπίσει επιστημονικά κριτήρια για του ενδοκρινικού διαταράκτε. Και να σας πω, να είμαι ευέλικτο. Αν υπάρχουν τεχνικοί λόγοι για να καθυστερήσει κανεί, δεν είχα κανένα πρόβλημα, αλλά είμαι αμήλικτο όταν οι λόγοι είναι πολιτικοί. Και αυτό δυστυχώ συμβαίνει αυτή τη στιγμή εδώ. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι και αυτή σαφέστατη. Η Κομισιόν θα έπρεπε να έχει θεσπίσει τα σχετικά κριτήρια, τα σχετικά επιστημονικά κριτήρια στον Δεκέμβριο του 2013 και διαβάζοντα από την απόφαση του δικαστηρίου δεν υπάρχει διάταξη του κανονισμού η οποία απαιτεί εκτίμηση επιπτώσεων. Δεν είμαι κατά τη εκτίμηση επιπτώσεων. Σαφώ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και σε αυτήν την περίπτωση. Όμω πριν καν ξεκινήσει μια τέτοια εκτίμηση, θα έπρεπε να είχαν θεσπιστεί επιστημονικά κριτήρια. Ήδη τον, τον Ιούλιο του 2013 αυτή ήταν έτοιμα, ήταν σε κάποια σιρτάρια του Μπερλεμόν, σκονίζονταν και θα έλεγα ας ξεσκονίζουμε τα σιρτάρια μας, ας τα ανοίξουμε και α κάνουμε αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε μόλις εντός ε, λίγων εβδομάδων. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια κυρία Ριβάση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. θα έλεγα ότι από τη στιγμή που οριστήκατε ως Επίτροπος Υγείας η ομάδα των Πρασίμων σας ενημέρωσε ότι ε, οι διαταράκτες, οι ενδοκρινικοί θα ήταν ένα από τα θέματα προτεραιότητας. Ε, αυτό ήταν το 2014. Το 2016 λοιπόν ε, ήρθε και δεν έγινε τίποτα. Η υπουργό Υγείας της Σουηδίας έφτασε στο Κοινοβούλιο, έφτασε μέχρι και το ε, Γενικό Δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο σας καταδίκασε χωρίς επιφύλαξη. Αυτή η καταδίκη του Σεπτεμβρίου λέει ότι η Κομισιόν δεν σεβάστηκε το ε, νόμο, αλλά ούτε και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποτε ε, σας ρωτάμε για αυτό το θέμα κρύβεστε πίσω από μία οικονομική ε, μελέτη επιπτώσεων η οποία δεν είναι απαραίτητη και ε, δεν δικαιολογεί το γεγονός ότι παραβιάσατε τις υποχρεώσεις σας. Κύριε Επίτροπε, λοιπόν, πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε μαζί αν η Κομισιόν δεν σέβεται το δίκαιο, τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι λοιπόν η εμπιστοσύνη που μπορεί να έχει ο τον άλλον. Μέσα στους επόμενους μήνες ε, πρέπει ταχαίως να δράσουμε για να μπορέσουμε να ορίσουμε τα στοιχεία για αυτούς τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Και ήδη έχουμε εδώ από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος ε, τα έγγραφα που δείχνουν τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί από αυτούς. Ακόμη και αύριο λοιπόν μπορείτε να τα έχετε στα χέρια σας και να τα θεσπίσετε. Δράστε λοιπόν γρήγορα. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταία συντάκτρια, η κυρία Κλόνεν. Έχετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύμφωνα με τον κανονισμό για τα βιοκτόνες ουσίες, ε, το 2013 η Κομισιόν ε, θα έπρεπε να έχει πράξεις ε, κατεξουσιοδότηση για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Αυτό δεν συνέφη. Η Κομισιόν δεν υιοθέτησε αυτές τις πράξεις κατεξουσιοδότηση και με αυτόν τον τρόπο δεν ε, τήρησε την υποχρέωση της, ε, την νομική της υποχρέωση να ε, λάβει μέτρα. Τον Ιούλιο του 2014 η Σουηδία κατέθεσε μια προσφυγή που υποστρέφθηκε από άλλα κράτη-μέλη και τη χώρα μου, τη Φιλανδία, στο δικαστήριο. Το δικαστήριο αποφάνθηκε το 2014, παρόλα αυτά η Κομισιόν διστάζει να εγκρίνει αυτές τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Γιατί λοιπόν δράσατε τόσο αργά. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που δείχνουν πως η Κομισιόν ε, διψάει για εξουσία και διψάει για πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Ε, ειδικά σε περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να το κάνει και τώρα που πρέπει δεν το κάνετε. Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Είναι μια σημαντική απειλή για τα έμβρια που ε, μπορεί να έχουν προβλήματα ε, στο μεταβολισμό τους ε, και να έχουμε και παραμορφώσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν τα επιστημονικά κριτήρια για να ορίσουμε τις ιδιότητε ε, της ε, διατάραξης ε, του μεταβολισμού. Πρέπει να έρθουμε στην Κομισιόν για να τις πάρουμε. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις τέθηκαν κύριε Επίτροπε και τώρα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία να αποσαφηνίσω τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, κατόπιν μιας ε, απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου ε, σε σχέση με την υπόθεση της Σουηδίας κατά της Επιτροπής για τους ενδιοκρινικούς διαταράκτες. Σήμερα θέλω να διασκορπίσω πάσα αμφιβολία σε σχέση με τις προθέσεις της Κομισιόν. Από ό,τι φαίνεται έχει υπάρξει κάποια παρεξήγηση να είμαι λοιπόν απολύτως σαφής. Η Κομισιόν έχει σταθερή πρόθεση να σεβαστεί την απόφαση του δικαστηρίου. Και θα το κάνουμε. Η απόφαση 16 Δεκεμβρίου 2015 αποφάνθηκε το δικαστήριο ότι η Κομισιόν παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς ε, δεν έθεσε συνεκτικά κριτήρια για να ε, καθορίσει τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και αυτό είναι αλήθεια. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, η Κομισιόν είχε αναλάβει μία σαφή δέσμευση με κατεξουσιοδότηση πράξη να θέσει τα κριτήρια μέχρι το Δεκέμβριο του 2013, πριν τρία χρόνια δηλαδή. Επίσης, το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν υπάρχει διάταξη σε αυτό τον κανονισμό που να απαιτεί τη διεξαγωγή μελέτης επιπτώσεων. Επίσης, από την πλευρά του δικαστηρίου είναι σαφέστατη η θέση αυτή, αλλά να συνεχίσω. Ξέρω ότι οι αντιδράσεις της Κομισιόν σε αυτή την απόφαση δέχτηκαν ε, κάποιες κριτικές και φυσικά σε μια δημοκρατία είναι κάτι λογικό. Επίσης η απόφαση σε σχέση με τη μελέτη αντικτύπων φυσβητήθηκε από κάποιους βουλευτές και διάβασα πολύ προσεκτικά τις επιστολές που εστάλθηκαν σε μένα ή στον πρόεδρο Γιούνκερ. Τις διάβασα πάρα πολύ προσεκτικά και έχω όλα αυτά τα έγγραφα στο γραφείο μου. Η Κομισιόν όμω θέλει να αποσαφηνίσει ότι η μελέτη αντικτύπου αποτελεί ένα χρήσιμο και ουσιαστικό εργαλείο για την καθοδήγηση των μελλοντικών αποφάσεων για τη θέσπιση κριτηρίων. Και συμφωνώ μαζί σα, λέτε, η μελέτη επιπτώσεων είναι ενδιαφέρον εργαλείο και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τέτοια κριτήρια. Ο ορισμός του ΠΟΗ δεν αρκεί. Και εσείς το είπατε ότι υπάρχουν διάφορες αποκλίνουσες θέσεις. Δεν είναι εύκολο να περιγράψει κανεί τα κριτήρια. Η Κομισιόν αποφάσισε το 2013 να διεξαγάγει μία μελέτη επιπτώσεων, όχι μόνο επειδή ήταν επιστημονικά πολύπλοκο το θέμα, αλλά και επειδή θα υπρόκειται για μία πρωτοποριακή δουλειά. Δεν υπάρχει πρώτερη νομοθεσία στον τομέα αυτό. Και όλοι το γνωρίζουμε ότι δεν διατίθεται. Καταρχήν, η επιστήμη δεν συμφωνεί για το πώς πρέπει να καθοριστούν αυτά τα επιστημονικά κριτήρια και μαζί έχουμε κάνει αυτές τις συζητήσεις. Υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις. Ακόμη υπάρχουν αυτές οι αποκλίνουσες απόψεις. Η επιστημονική κοινότητα διαφωνεί σε σχέση με το πώς θα πρέπει να προσδιοριστούν οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, γιατί πρέπει να μιλήσουμε εδώ για κανονιστικά ζητήματα. Επίσης, μπορούμε αυτά τα επιστημονικά κριτήρια να τα θέσουμε σε ένα κανονιστικό πλαίσιο. δεν υπάρχουν δεσμευτικά κριτήρια σε τρίτες χώρες για να εντοπιστούν οι χημικές ουσίες ενδοκρινικών διαταρακτών. Επίσης, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορισμένα κράτη-μέλη υποστηρίζουν μία ε, προσέγγιση που να οφείλεται στην πρόληψη, ενώ άλλα που να οφείλεται στον κίνδυνο, που να βασίζεται στον κίνδυνο. Και κάναμε αυτή τη μελέτη δικτύπων για να διευκολυνθούμε. Και εδώ συμπεριλαμβάνω και σας ως μέλη του Κοινοβουλίου Δηλαδή δεν πρέπει να ενημερωθείτε για να πάρετε μία σωστή απόφαση. Η Κομισιόν γνωρίζει πλήρως ότι έχει λήξει η προθεσμία, έχει εκπνεύσει η προθεσμία και έχει κάθε πρόταση να σεβαστεί την απόφαση του δικαστηρίου. Αναμφισβήτητα, η προετοιμασία της μελέτης συντικτύπου έχει προχωρήσει πολύ και σε απάντηση της απόφασης του δικαστηρίου Κομισιόν πριν από το καλοκαίρι το 2016 θα παρουσιάσει νέα επιστημονικά κριτήρια για τους ενδιοκρινικούς διαταράκτες. Όπως γνωρίζετε, θα πρέπει να παρουσιάσουμε δύο διαφορετικές πράξεις. Πρώτον, εφαρμοστικό κανονισμό που να περιλαμβάνει τα κριτήρια που θα εφαρμόζονται στις χημικές ουσίες που εμπίπτουν ε, στον κανονισμό της φυτοπροστασίας και την λεγόμενη διαδικασία της πράγας και δεύτερον κατεξουσιοδότηση πράξης που να περιλαμβάνουν κριτήρια που να εφαρμόζονται δυνάμει του κανονισμού, των κανονισμών για τα βιοκτώνα. Διασφαλίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δεσμεύεται η Κομισιόν να σεβαστεί την απόφαση του δικαστηρίου. Επομένως, πριν από το καλοκαίρι θα παρουσιάσουμε κριτήρια τα οποία θα είναι προσδιορισμένα με αντικειμενικό τρόπο και θα βασίζονται σε επιστημονικές αποδείξεις. Εδώ ο δικαστής έχει διαφορετική άποψη όμως πρέπει να κατανοήσετε σήμερα ότι θέλουμε να δούμε περισσότερες συγκλίνουσες απόψεις. Η νομοθεσία μας σε αυτούς τους δύο τομείς ε, θεωρείται μεταξύ των πιο αυστηρών στον κόσμο και θέλω να διασφαλίσω ότι είναι υψηλό επίπεδο προστασίας για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες θα διατηρηθεί πλήρως. Τα ενδιάμεσα κριτήρια για το να ε, διαπιστώσουμε, να βρούμε τους ενδοκρινικούς διαταράκτες είναι νομικά δεσμευτικά και εφαρμόζονται. Φυσικά όλα αυτά δεν αρκούν θα πρέπει άμεσα μέχρι αυτό το καλοκαίρι να καθορίσουμε συνεκτικά κριτήρια για τους ενδοκρινικούς διεκτεράκτες. Εγώ συχνά σας ενημέρωνα για αυτό το πολύπλοκο ζήτημα. Ακολουθήσαμε μια πολύ διαφανή διαδικασία και αυτό σκοπεύω να κάνω. Θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού έτσι ώστε να καταλήξουμε στο να λάβουμε την καλύτερη απόφαση για αυτό το σημαντικό θέμα. Και θα ήθελα να έχω επικοδομητική υποστήριξη από εσά για τα βήματα που θα κάνουμε στο εγγύ μέλλον. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και τώρα ο λόγος στου επιμέρου ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Γκίζεκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη Επίτροπε Ανδρουκαίτη, αγαπητοί συνάδελφοι, χρειαζόμαστε έναν ορισμό για Αυτές τις ουσίες που ονομάζονται ενδοκρινικοί διαταράκτες είναι ένα νομικό δικαίωμα και υποχρέωση υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών. Μας μιλάει η Κομισιόν με τεχνικούς όρους για επιστημονικά ζητήματα που έχουν επιστημονική ευθύνη. Όμως, το 2015 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ορίζει ε, στην απόφασή του ότι η Κομισιόν παρέλειψε μια προθεσμία. Αυτό που ε, έκανε ξεκάθαρο εδώ και μήνες το ΕΛΚ ε, ισχύει λοιπόν. Πρέπει η Κομισιόν άμεσα να θεσπίσει τα κριτήρια και αν ε, το καταφέρετε αυτό μέσα στο 2016 θα έχετε κάνει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν βάσει της απόφασης του δικαστηρίου υπάρχει αυτή η παραβίαση των υποχρεώσεων, ε, πραγματικά η Κομισιόν πρέπει να απαντήσει για ποιο λόγο συνέβη αυτό. Είπαν ότι υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση. Φαίνεται ότι ε, υπάρχουν πάρα, πάρα πολλά δεδομένα που πρέπει να συλλέξουμε σε επιστημονικό επίπεδο και η Κομισιόν, από ό,τι καταλάβαμε, είναι σε καλό δρόμο και ε, από τη δική μου ομάδα, το ΕΛΚ, θα έχει υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο Πότς, ένα Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, εδώ και πέντε χρόνια συζητάμε αυτό το ζήτημα και οι Ευρωπαίοι έχουν εκτεθεί όλο αυτό το διάστημα σε ουσίες που οδηγούν σε καρκίνο, ψυχικές ε, νόσους, ε, έλλειψη γονιμότητας κτλ. Έχουμε ε, συζητήσει γι' αυτό το θέμα με πολλές προεδρίες. Η Ολλανδική Προεδρία έθεσε αυτό το θέμα ως προτεραιότητα της, αλλά δεν είναι καν εδώ. Κύριε Επίτροπε, μιλήσαμε για αυτό το θέμα και υποσχεθήκατε ότι θα τηρήσετε κανόνες που δεν τηρήσατε. Σήμερα πρέπει να οδηγηθούμε σε μια γρήγορη ρύθμιση και είπατε πως οι επιστήμονες δεν συμφωνούν σε αυτό το θέμα. Η Κομισιόν ως τώρα δεν αποδέχτηκε την απόφαση του δικαστηρίου και δεν ε, θέσπισε τα κριτήρια. Ποιος είναι ο λόγος που η Κομισιόν εδώ και χρόνια δεν ε, ε, λαμβάνει υπόψη της ούτε τους πολίτες, ούτε το δικαστήριο, ούτε το κοινοβούλιο. Είναι δική σας ευθύνη αυτό. Έχει να κάνει με τις διαπραγματεύσεις για την TTIP. Ε, επειδή αυτός ο ορισμός ε, δεν θα βοηθούσε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ποιος είναι ο λόγος ε, που δεν συμμορφωνόσαστε με την απόφαση του δικαστηρίου. Θέλουμε πραγματικά αυτή τη στιγμή να έχουμε αυτή, αυτό τον ορισμό. Θα μας τον δώσετε, είπατε. Ευχαριστούμε. Όμως, τι γίνεται με την εμπιστοσύνη των πολιτών ε, στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Αυτό ε, δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Πρόεδρος, όντως είναι σημαντικό το θέμα. Αλλά παρακαλώ να τηρείτε όλοι το χρόνο σας. ε, εκ, λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε ε, Πίτρο Πέδρο Καΐτης εδώ και χρόνια. Ε, ε μιλάμε για λιπάσματα, για τα πλαστικά, ε, για όλα αυτά τα προϊόντα που περιλαμβάνουν αυτούς τους διαταράκτες. Ακόμα και σε μικρή δόση προκαλούν προβλήματα στους ανθρώπους και στα ζώα, όπως ας πούμε καρκίνο και άλλες ασθένειες. Αυτό έχει να κάνει με τη χρήση αυτών των χημικών οι ε, κίνδυνοι από τους ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες δεν είναι κάτι καινούριο. Τι κάνει όμως ε, η Κομισιόν έχει παραλείψει να τηρήσει μια προθεσμία και ξεκάθαρα ξεχνάει να κάνει το καθήκον της ενώ εμείς καθημερινά και μέρα με τη μέρα έχουμε όλο και μεγαλύτερη επιβάρυνση από αυτούς τους διαταράκτες. Ε, γιατί αναλαμβάνουμε αυτό τον κίνδυνο. Ε, ήρθε η στιγμή οι πολίτες της Ευρώπης να προστατευτούν από αυτές τις ουσίες. Αυτό περιμένουν ακριβώς από εμάς. Γι' αυτό μας εξέλεξαν εδώ σε αυτό το σώμα και ε, δεν πρέπει να εκπροσωπούμε κανέναν, ούτε τη φαρμακευτική βιομηχανία, ούτε κανέναν άλλον. Ευχαριστώ, ο κύριος Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, Ευχαριστώ. Ξεκινήσατε πολύ ωραία λέγοντας ότι θα συμμορφωθείτε με την απόφαση του δικαστηρίου και με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και μετά άρχισαν οι οριστείες γύρω από την εκτίμηση επιπτώσεων. Τα πράγματα είναι απλά. Το δικαστήριο είπε τα επιστημονικά κριτήρια είναι τα μόνα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν. Ήταν σαφές το 2013 και είναι και σήμερα αφού ήταν έτοιμα το 2013, γιατί δεν δημοσιεύονται σήμερα. Είμαστε στο 2016. Γιατί, μήπως θέλετε να περιμένετε πράγματι για την περίφημη εκτίμηση επιπτώσεων για να καταστρατηγήσετε εν τέλει την απόφαση. Γιατί η απόφαση λέει σαφέστατα ότι το εγχείρημα είναι απολύτως επιστημονικό. Αν θέλετε λοιπόν να καταστρατηγήσετε την απόφαση του δικαστηρίου, αυτό είναι ντροπή. Πρόεδρος, ο επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Εύη. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρα. Κύριε Πίτροπε, η απόφαση του δικαστηρίου αναγνώρισε ότι η Κομισιόν έχει καθυστερήσει στο να θεσπίσει τα κριτήρια για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Η καθυστέρηση αιτιολογείται με την αναγκαιότητα να γίνει μια αξιολόγηση κόστους ωφέλους. Βέβαια αυτό είναι αμφισβητήσιμο καθώς τα κριτήρια επιστημονικής αξιολόγησης δεν μπορούν να ακολουθούν τις εμπορικές απαιτήσει. Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε το Μάρτιο του 2015 εκτίμησε το κόστος το ετήσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω στην έκθεση στους δικρονικούς διαταράκτες ε, ε, περίπου στο 360 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό οφείλεται στο ε, ότι δυστυχώς κάθε χρόνο πληρώνουμε, τα πληρώνουν αυτό το κόστος 60.000 νεογέννητα ε, που εκτίθενται σε αυτές ε, τις ουσίες ε, και παρουσιάζουν προβλήματα. Πρόκειται για μωρά τα οποία έχουμε στερήσει το μέλλον τους. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνω το πρώτος γύρος των ομιλητών και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκροστέτ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζεται για ένα τόσο σοβαρό θέμα να κάνουμε του αντικοινωνικού διακτάκτε ε, ενώ εμείς κούρσαμε τον κόσμο του κινδύνου εδώ και πολύ καιρό. λέτε αντικτύπου, ναι, ε, πολύ ωραία, αλλά θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα και θα έπρεπε ήδη να την έχουμε στη διάθεσή μας. Εμείς τι ζητάμε την, ε, τη θέσμηση κριτηρίων για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες βάσει επιστημονικών μελετών. Εμείς Αναρωτηθήκαμε από ποιο σημείο και μετά υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία. Πρέπει να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Βέβαια, η βιομηχανία θα πρέπει να βρει εναλλακτικέ λύσεις και εδώ μπορούμε να φανταστούμε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην πίεση ορισμένων λόμπι. Αυτό είναι θλιβερό. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μιλά για το ευνομοθετήν, σήμερα ε, για ένα θέμα στο οποίο θα έπρεπε να φέρει προσθέμενη αξία στο θέμα της δημόσιας υγείας, ε, πώς θα το κάνει αυτό θα πρέπει να προτείνει νομοθεσία για το θέμα αυτό. Καθυστερήσατε, μα, συγγνώμη, κερδίσατε 30 δευτερόλεπτα. Τώρα ο κύριος Σπαρνιό για μισή λεπτό. Είναι σκάνδαλο. Είναι πολιτικό σκάνδαλο. Αυτό έχουμε μπροστά μας. Όντως, η απόφαση του δικαστηρίου λέει ότι πρέπει να κάνουμε γρήγορα δεν είναι τεχνικό το πρόβλημα. Είναι καταρχάς ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας, της υγείας των ανθρώπων. Ευρωπαίοι πεθαίνουν κάθε μέρα από καρκίνους εξαιτία των παρασιτοκτόνων, για παράδειγμα, που είναι προϊόντα που αποτελούν διαταράκτες. Οι συσκευασίες παιδικών παιχνιδιών, απλά εισιτήρια τα οποία περιέχουν ακριβώς ενδοκρινικούς διαταράκτες. Το θέμα είναι λοιπόν να υπερμενθούμε τη υγείας των Ευρωπαίων, ανδρών και γυναικών. Έτσι ώστε οι δυσπλασίες, οι καρκίνοι, αλλά και άλλου είδους επιπτώσεις δεν πλήττουν την υγεία μας. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε. Βεβαίως είναι οικονομικό το πρόβλημα. Ε, κάποιοι αναφέρθηκαν σε αυτό. Πόσο κοστίζει. Να σας πω ότι κοστίζει 1,3 του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, το σύνολο των βλαβών, στην υγεία. Λόγω ακριβώ ενδοκρινικών διαταρακτών. Αυτό είναι το κόστος. Και αυτό λοιπόν λέει και η απόφαση του δικαστηρίου. Το δικαστήριο δεν είπε ότι πρέπει να ξεκινήσετε να κάνετε μια μελέτη επιπτώσεων κλπ. Όχι. Το είπαν και οι προλαλήσεντες επιστημονικά κριτήρια για να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ευχαριστώ, κύριε Άουχεν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ πίτροπε. Είναι ένα πολλαπλό σκάνδαλο. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν συμφωνούν οι επιστήμονες για τα επιστημονικά στοιχεία. Στη Δανία υπάρχει μια δελεχής μελέτη, η οποία έχει δημοσιευθεί σε όλη την Ευρώπη και μιλά για ε, την επιρροή στον εγκέφαλο των αγέννητων παιδιών. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις ακόμα και στη γονιμότητα των γυναικών, των ανδρών, συγγνώμη. Αυτό που ακόμα δεν έχουμε ε, δει είναι κατά πόσο θα, πληχθεί, θα πληγεί η βιομηχανία εάν δεν αναλάβει δράση και δεν βρει εναλλακτικέ λύσεις. Αν δεν θεσπίσουμε κριτήρια, οι εταιρείε δεν θα μπορέσουν να κάνουν σταδιακή απομάκρυνση αυτών των ουσιών και να βρουν εναλλακτικέ λύσεις. Πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε τόση προσπάθεια για να ικανοποιήσουμε την παραδοσιακή βιομηχανία. Τώρα ο λόγος του κύριο Μπάλετ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να επαναλάβω ότι οι ενδοκρινικοί διαταράκτες ε, είναι πηγή μεγάλης αβεβαιότητας και ανησυχία, όχι μόνο εδώ, αλλά εδώ στο Κοινοβούλιο δηλαδή, αλλά και στο μυαλό των πολιτών, υπάρχουν παντού τις συσκευασίες, στα ενδύματα. Πρέπει λοιπόν να ε, βρούμε ξεκάθαρα επιστημονικά στοιχεία και χαίρομαι ιδιαίτερα που λέτε ότι πολύ σύντομα πριν το καλοκαίρι θα μπορέσετε να έχετε την μελέτη επιπτώσεων. Είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε επικοινωνία σε ευρία βάση. Ακούγεται σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Βέβαια υπάρχουν ήδη κάποιοι αυστηροί κανόνες για τη χρήση χημικών, στα πλαστικά, στα παιχνίδια. Έχουμε τους κανόνες ε, βάσει της οδηγίας REACH. Υπάρχουν κάποιες διατάξεις εκεί για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, όμως τώρα ήρθε η στιγμή να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και υπόθηκε ξεκάθαρα πρέπει να υπάρχει μέγιστη προστασία των καταναλωτών. Πρέπει να δράσουμε έτσι ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον ώστε να βρεθούν και εναλλακτικέ. Ευχαριστώ. Η κυρία... Κύριε Σαρβού. Κυρία Πρόεδρε, οι διαταράκτες είναι παντού και είναι πολύ επικίνδυνοι. Βρίσκονται στα παιχνίδια, σε καλλιντικά και αποτελούν κίνδυνο για την υγεία. Πρέπει λοιπόν να αποτελέσουν ένα αντικείμενο ρύθμισης. Τα κριτήρια, τα σχετικά κριτήρια, πρέπει να είναι επιστημονικά και να μην έχουν σχέση με τις οικονομικές πτυχές. Η Κομισιόν όταν ήρθε η ώρα να θεσπίσει τα κριτήρια αυτά, ασχολήθηκε πιο πολύ με την οικονομική πτυχή παρά με την υγεία. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας. Χρειαζόμαστε λύση σήμερα. Δεν νομίζω ότι η Κομισιόν έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη ανάληψης ταχείας δράσης. Το αντίθετο. Πρώτον ανέβαλε τη λήψη μέτρων για ένα χρόνο, και φοβούμαι ότι έχει χάσει τι προτεραιότητε της. Πρόεδρο, ο κύριο Στά, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η εκτίμηση επιπτώσεων και όλη αυτή η ιστορία έχουν σχέση με τα λόμπι, φοβούμαι. η βιομηχανία φοβούμε θέλει να παρισφρήσουν άλλα κριτήρια στη συζήτηση. Φοβούμε δηλαδή ότι θα καταλήξουμε υπό την πίεση της βιομηχανίας να κάνουμε κάτι μόνο για τους πιο προβληματικούς διταράκτες. Έχω εδώ δύο ποτά. Το ένα περιέχει 40% το αλκοόλ, το άλλο 3. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει αλκοόλ στην πύρα, να υπάρχει στο απόσταμα. Αυτό προσπαθεί να κάνει βιομηχανία. Μα πείσει ότι το ένα είναι διαταράξη και το άλλο δεν είναι. Λοιπόν, σα προειδοποιώ. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να θεσπιστούν τα κριτήρια. Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής, ο κ. Μπουσόη. Παρακαλώ. Αγαπητέ πίτροπε η παρουσία των κρινικών διαταρτών στο περιβάλλον προκάλεσε ανησυχίε τα τελευταία χρόνια γιατί παρατηρήσαμε επιβλαβή αποτελέσματα στην αναπαραγωγή ε, και στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες ε, αποτελούν μια πρόκληση καθώς τα αποτελέσματα εξαρτώνται από το μέγεθος αλλά και το χρόνο της έκθεσης. Ορισμένοι από τους συναδέλφους μου και είμαι πεπισμένος ε, ότι θέλουν να προστατεύσουν την υγεία των πολιτών ε, κατά των ειδοκρινικών διαταρακτών ε, με τον καλύτερο τρόπο. Άσκησαν σκληρή κριτική στην Κομισιόν, αλλά πιστεύω ότι παρά την απόφαση του δικαστηρίου, η αρχική πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τη μελέτη επιπτώσεων ήταν ο καλύτερος τρόπος για να καταλήξει στη θέσπιση αναλογικών και επιστημονικών κριτηρίων. Συνεχίζεται η διαδικασία και καλωσορίζω την αποφασιστικότητα του Επιτρόπου Ανδρουκαϊτής που τοποθετήθηκε εδώ και είπε ότι θα επιταχύνει τη διαδικασία. Τώρα δεν υπάρχει νομικό κενό, προστατεύονται οι πολίτες από την φυστάμενη νομοθεσία, από το ΡΙΤΣ, από τον κανονισμό για τα βιοκτώνα. Αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμόζεται και επικαιροποιείται με τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία. Ο στόχος τελικά είναι να καθοριστούν κριτήρια που θα μπορούν να εντοπίσουν καλύτερα τι ουσίε που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε ρεαλιστικές συνθήκες. Αυτό μας επιτρέπει να αποφασίσουμε τι θα απαγορεύσουμε ή σε ποιες ουσίες θα απαγορεύσουμε τη χρήση τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε εδώ κάποια τεχνική υποστήριξη. Να σβήσει κάποιος το μικρόφωνο του κύριου Στάς, παρακαλώ. γιατί αν συνεχίσει να είναι ενωμένο προκαλεί θόρυβο. Λοιπόν, η κυρία Ριβάση θα ήθελε να σας θέσει μια ερώτηση με μπλε κάρτα, αν δέχεστε, κύριε Μπουσόη. Κύριε Μπουσόη, λέτε, πρέπει να εξαλείψουμε τους μικρούς διαταράκτες στο όσο το περισσότερο δυνατόν γιατί θέτουν προβλήματα. όμω το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει δόση, δεν υπάρχει κατόφλι. Σε ένα πολύ μικρό επίπεδο μπορεί επίσης να έχουν πολύ σημαντικές συνέπειες. Γι' αυτό πρέπει να τους διορίσουμε έτσι ώστε να εξελιχθούν. Δηλαδή δεν αρκεί εδώ να πούμε θα τους εξελίψουμε όσο δυνατό περισσότερο. Εάν υπάρχουν θα πρέπει να τους αφαιρέσουμε. Και θα πρέπει να πούμε στη βιομηχανία, έχετε δύο χρόνια για να βρείτε μια λύση. Κύριε Μπουσόη. Συμφωνώ μαζί σας. Το ίδιο λέω κι εγώ. Αλλά κατάλαβα και την αρχική πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διεξαγάγει μια μελέτη για να δει ποια ακριβώς είναι τα πιο σαφή κριτήρια. Γιατί αν δεν έχουμε κριτήρια που να υποστηρίζει και η επιστημονική κοινότητα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσδιορίσουμε σωστά τα κριτήρια. Πρόεδρος, ευχαριστώ για την απάντησή σας. Ο κύριος Καπούτο τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η Κομισιόν ε, καθώς ε, δεν προέβησε κατοξιδόξη πράξης ε, για την θέσπιση κριτηρίων για τους οδικρινικούς διαταράκτες δεν σεβάστηκε τις υποχρεώσεις της βάσει του κανονισμού για τα βιοκτώνα επίσης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, κατόπιν ε, προσφυγής της Σουηδίας ενώ γνώρισε παραβίαση του δικαίου από την πλευρά της Κομισιόν με αυτή την καθυστέρηση από το Σεπτέμβριο του 2013 μας δείχνει η Επιτροπή ότι δεν μπορεί να, απαιτεί, να απαντήσει στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων πολιτών για προστασία της υγείας. Ε, φτάνουν οι δικαιολογίες για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και φτάνει και η αναμονή για τη μελέτη αντικτύπου. Εμείς περιμένουμε την ταχύη υιοθέτηση μέτρων που να οδηγούν στη θέσπιση επιστημονικών κριτηρίων για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλίσει των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Χόισλινγκ, σε ένα λεπτό. Κύριε ε, Επίτροπε, η πίστη των ε, πολιτών στη δική μας πολιτική έχει ε, πραγματικά υποσκαφθεί και αυτό είναι σκάνδαλο. Εγώ είμαι αγρότης και δεν έχω καμία κατανόηση να ε, έχουμε στα λοιπάσματα έλλειψη αξιολόγησης της ύπαρξης ενδοκρινικών διαταρακτών. Έχουμε προβλήματα στους χρήστες και στο περιβάλλον και στους καταναλωτές. Δεν νομίζω ότι είναι παρεξήγηση όπως είπατε. Έγινε συγκεκριμένη παρέμβαση από το λόμπι της ε, γεωργικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας ε, που φοβάται ότι θα χάσει έσοδα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να λάβετε πιο σοβαρά υπόψη σας τα συμφέροντα των καταναλωτών και ε, ε, επίσης στα καλλιντικά θα πρέπει να δούμε πώς θα, τι θα γίνει με τα κριτήρια και εκεί πρέπει να αναλάβουμε δράση. Ευχαριστούμε πολύ. κύριος Άρημον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Πολλά από τα αντικείμενα της, από τα αντικείμενα της καθημερινής μας ζωής περιλαμβάνουν ενδοκρινικούς διαταράκτες ας πούμε ε, τα ξύλα που έχουν ε, ε, από πάνω λούστρο, τα, τα πλαστικά, τα παιχνίδια που έχουν τα παιδιά, ακόμα και αυτά που παίρνουν στο σχολείο τα εξαρτήματα. Όλα αυτά οδηγούν σε καρκίνο, σε διαβήτη, σε υπογονιμότητα. Χρειάζεται λοιπόν άμεσα δράση. Τον ε, Δεκέμβρη ε, η Κομισιόν παρέλειψε να συμμορφωθεί με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και μίλα ε, για έλλειψη επιστημονικών κριτηρίων. Στην ουσία αυτές οι επικίνδυνες ουσίες πρέπει να ρυθμιστούν αυστηρά Αυτές οι ουσίες είναι ξεκάθαρα επιβλαβείς και έχουν και σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνία. Υπάρχουν κάποιες μελέτες οικονομικές που αναφέρουν ότι αυτές οι ασθένειες επιβαρύνουν τα ταμεία μας με 60 δις ευρώ. Ε, έτσι λοιπόν θα πρέπει κάτι να κάνετε για να προστατέψετε καλύτερα την υγεία των πολιτών. Είναι η αρχή της πρόληψης. Ακόμα και αν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία ότι μία ουσία ε, είναι επιβλαβής ή όχι, θα πρέπει αν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία για το πόσο επιβλαβής είναι μία ουσία, θα πρέπει αυτή η ουσία να μην βρίσκεται στην Ευρώπη γιατί πρέπει να προστατεύουμε τους πολίτες και όχι τους μεγάλους ομίλους. Αυτοί πρέπει να βρουν εναλλακτικέ. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Μπορζάν. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με την απόφαση του δικαστηρίου. Είναι προφανές ότι η Κομισιόν δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις της που έχουν σχέση με την υγεία των πολιτών. Οι ουσίες αυτές επηρεάζουν τα μάλλα την υγεία μας. Επηρεάζουν τις ορμόνες μας. Και μάλιστα οι ουσίες αυτές βρίσκονται σε συσκευασίες, τα πλαστικά, παντού. Όσον αφορά τους ενδοκρινικούς διθαράκτες υπάρχουν διάφορες και διαφορετικές θεωρίες. Μερικές μπορεί να μην είναι ακριβής. Όμως η απόφαση του δικαστηρίου είναι εκεί και δυστυχώς διακυβεύεται εδώ το κύρος της Κομισιόν. Καλό την Κομισιόν να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την απόφαση του δικαστηρίου και να θεσπίσει κριτήρια για τους ενδοκρινικούς διταράκτες. Επιστημονικά κριτήρια, ρεαλιστικά και καλά για την υγεία. Πρόεδρος, και τώρα Άντερσον, ευχαριστώ πολύ. Οι διδαράκτες προξενούν βλάβες έμβρια, προξενούν καρκίνους. Τα μικρά παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Επηρεάζει τον εγκεφαλός τους και η αναπτυξή του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει ευθύνη να προστατεύσει τους πολίτες κατά των ενδοκρινικών διαταρακτών. Και όμως η Επιτροπή παίζει καθυστερήσεις, κολυσιεργεί έφτασε στο σημείο να καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να δείτε τα πράγματα σοβαρά, κύριοι τη Κομισιόν, και να μην προστατεύετε τα συμφέροντα τη βιομηχανία. Πρόεδρο. Και τώρα, Πέτερλε. Παρακαλώ, ένα μισή λεπτό. Κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο προστάτης η καρκίνη, οι διαβήτες, τα καρδιαγγειακά όλες αυτές οι νόσοι οι προβλήματα αναπαραγωγής, γονιμότητας και όλα αυτά γνωρίζουν τρομακτική αύξηση και έχουμε χημικές ουσίες όπως το PBA, PB, PD, ε, παρασιτοκτόνα και άλλα φυτοπροστατευτικά τα οποία αποτελούν σημαντικό πρόβλημα. Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες δίνονται να προκαλέσουν μη αντιστρεπτά αποτελέσματα. Το κόστος κατέτος ξεπερνά, εκτιμάται, τα 150 δισεκατομμύρια. Ας προστατεύσουμε λοιπόν τις πλέον ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και δει τις ε, εγγύους, τα νεογνά τα μωρά. Η πρώτη μας προτεραιότητα λοιπόν πρέπει να είναι να προστατεύσουμε την υγεία του πληθυσμού. Στον τομέα της υγείας, που είναι μία από τις τρεις βασικές μας προτεραιότητες, πρέπει να έρθουμε πιο κοντά στους πολίτες μας. Πρέπει λοιπόν οι ενδοκρινικοί διαταράκτες να είναι στο κέντρο της πολιτικής μας πρόληψης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καλντεμόζο, παρακαλώ. Κυρία, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ πολύ. Καρκίνος, ε, οι δυσπλασίες, ε, ε, αποβολές εμβρίων κτλ. Έχουμε ένα μακρύ κατάλογο βλαβών που προκαλούνται από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Πρέπει λοιπόν να ευχαριστήσουμε τη Σουηδία που προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να αποσυφενήσει το θέμα αυτό και να αποκαλυφθεί ότι η Κομισιόν καθυστερεί για το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι αποδεκτό. Ξέρω ότι είναι πολύπλοκο το ζήτημα, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για τη μη ανάληψη δράσης για την προστασία της υγείας των πολιτών. Πολλοί με ρωτούν γιατί η Κομισιόν δεν ανέλαβε δράση και εγώ απαντώ δεν γνωρίζω και πραγματικά αυτό είναι ντροπιαστικό. Δεν αυξάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και α είμαστε ειλικρινεί, όσο καθυστερεί η Κομισιόν, τόσο πιο πολύ ευθύνεται για τι βλάβε στην υγεία των πολιτών. Σα παρακαλώ, καθορίστε κάποια κριτήρια τώρα, όχι αύριο. Κυρία Πιετικάνεν. Κυρία Πρόεδρε, οι διοκρινικοί διαταράκτες πλήττουν ε, όχι μόνο την υγεία της σημερινής γενιάς, ε, αλλά και των επόμενων γενεών. Πολλές φορές ε, οι συνέπειες εμφανίζονται μόνο στην επόμενη γενιά. Γι' αυτό μας πιέζει ο χρόνος. Υπάρχει ευρεία συνένεση σε σχέση με τη θέσπιση των κριτηρίων για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και το πώς θα μετρήσουμε τον αντίκτυπό τους. Δεν υπάρχει έλλειψη κριτηρίων. Έχουμε και τους κανονισμούς για τα βιοκτώνα, τον κανονισμό για το ρίτς. όλα αυτά αριθμίζουν την παρουσία αυτών των ουσιών στα ρούχα, στα χρώματα και αλλού. Και τώρα αποφασίστηκε ότι δεν χρειάζεται μελέτη αντικτύπου, γιατί εδώ τίθεται θέμα επιβίωσης, υγείας των ανθρώπων. Δεν πρέπει να έχουμε ως ε, πρώτο κριτήριο το οικονομικό. Θα πρέπει λοιπόν σε κάθε περίπτωση να σεβαστούμε τις απαιτήσει και το ελάχιστο που μπορούμε να περιμένουμε από την Κομισιόν είναι να ακολουθήσει αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές του δικαστηρίου. Και εγώ δεν θέλω να δεκτώ τώρα εδώ ότι διακυβεύεται η απόφαση να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών. Η κυρία Ρουής είναι ακατανόητη η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, μπορούμε να πούμε ότι εδώ και 20 χρόνια γνωρίζουμε ε, τις επιβλαβείς συνέπειες των ενδοκρινικών διαταρακτών για τη δημόσια υγεία και μάλιστα φτάσαμε σήμερα πρέπει να παρέμβει η δικαιοσύνη για να σας πει ότι ε, δεν υπάρχει πλέον λόγος να καθυστερείτε ούτε να εφευρίσκετε μελέτες αντικτύπου προκειμένου να θεσπίσετε τα κριτήρια για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Σας το είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι πάνω από τα οικονομικά συμφέροντα πρέπει να θέσουμε την υγεία των πολιτών. Και τώρα μας είπατε ότι θα έχουμε τα επιστημονικά κριτήρια το καλοκαίρι. Εγώ ελπίζω πράγματι να συμβεί αυτό και θα ήθελα να υπερισχύσει το κριτήριο της δημόσιας υγείας από ε, στο οικονομικό κριτήριο που ό,τι φαίνεται έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδρομή της θέσπισης των κριτηρίων. Σας ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώσαμε τις ε, συνεισφορές ε, των βουλευτών. Περνάμε τώρα στο Catch the Eye. Η κυρία Ζαμπόσκα πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Γενικά θεωρώ ότι είναι σωστό ε, η Κομισιόν εκ των προτέρων να προσπαθεί να εκτιμά το οικονομικό και κοινωνικό κόστος της έγκρισης και υιοθέτηση νέας νομοθεσίας. Όμως θα περίμενα η Κομισιόν πρώτα απ' όλα να ρυθμίζει το θέμα της ανθρώπινης υγείας. Τελικά έχει επιβεβαιωθεί η υποψία ότι οι ενδοκρινικοί διαταράκτες ε, μειώνουν τη γονιμότητα και των νυχτήρων και των ανθρώπων και ε, φαίνεται ότι η επένδυση σε συστήματα φιλτραρίσματος ε, και η διασφάλιση της πάταξης της μόλυνσης είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν από τα κράτη-μέλη. Φαίνεται ότι η χρήση αυτών των ουσιών στη γεωργία, στην κτηνοτροφία ε, είναι κάτι που χρησιμοποιείται ευρέως. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συζητούμε για την αύξηση των ενδοκρινικών διαταραχών και ασθενειών που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες είναι χημικέ ουσίε, οι οποίε μιμούνται τι ορμόνε και παρεμβαίνουν στο ορμονικό σύστημα με αποτέλεσμα να προκαλούν διαταραχέ στη γονιμότητα νέοπλασίε και διάφορε μορφέ καρκίνου. οι συγκεκριμένε ουσίε βρίσκονται όπω υπόθηκε σε πολλά προϊόντα καθημερινή χρήση, και ο μεμονωμένο καταναλωτή είναι αδύνατο να γνωρίζει την ύπαρξή του, αφού μάλιστα συχνά τα ίδια αυτά δεν φέρουν δήλωση περιεχομένου. Επομένω, είναι αναγκαίο η ευρωπαϊκή ένωση να επανεξετάσει την υπάρχουσα σχετική νομοθεσία και να υπάρξουν περισσότερε απαιτήσει σχετικά με τι χημικέ ουσίε που περιλαμβάνονται σε προϊόντα όπω τα τρόφιμα. επιπλέον θα πρέπει να γίνουν αλλαγέ όσον αφορά την αξιολόγηση την αδειοδότηση και του περιορισμού των ουσιών αυτών στα παραπάνω προϊόντα καθώ και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στον καθορισμό του κατά πόσο μια ουσία εν προκειμένου έχει τι ιδιότητε που πρέπει να απαγορευτούν. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, η, η κυρία... Ευχαριστώ. Ο Δεκέμβριος ε, του 2014 ε, είναι μια βαριά ημέρα για την Κομισιόν γιατί δεν τήρησε τις υποχρεώσεις της έναντι της δικαιοσύνης, έναντι των συνθήκων. Όμως είναι πολύ σκερός που η επιστημονική κοινότητα και το κοινοβούλιο την, ε, ε, εφιστούν την προσοχή για τα προβλήματα που δημιουργούνται στην υγεία. Ακριβώς αυτοί οι ενδοκρινικοί διαταράκτες είναι που δεν ε, είχαν τα αντικειμενικά κριτήρια, δεν είχαν θεσπιστεί κριτήρια για αυτούς ε, ήδη από το 2006 συζητούμε και εδώ και τρία χρόνια η Κομισιόν έχει την υποχρέωση να θεσπίσει τα κριτήρια. Είπατε ότι έχετε την ε, πρόθεση να συμμορφωθείτε πριν το καλοκαίρι. Το σημειώνουμε, όμως θα είμαστε και σε επαγρύπνηση για να ε, έχουμε... να δούμε ότι θα συμβεί. Ελπίζουμε να έχουμε λόγο να σας εμπιστευτούμε κύριε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κρύβεται και ουσιαστικά φιβρίστηκε ολογίες επειδή δεν έκανε αυτό που υποχρεούται να παρουσιάσει μέχρι το Δεκέμβριο του 2013 κριτήρια για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, ε, ουσίες που παρεμβαίνουν στο ορμονικό σύστημα του ανθρώπου και μπορούν να προκαλέσουν βαριές ασθένειες ε, και αναφερθήκατε σε ε, μία έλλειψη επιστημονικών στοιχείων για να μην κάνετε τίποτα και ουσιαστικά άλλα ενδιαφέροντα, οικονομικά ενδιαφέροντα από την χημική βιομηχανία σας επηρέασαν και φυσικά και η καθυστέρηση αυτή τη μελέτη αντικτύπου που έρχεται να το επιληθεύσει αυτό. Είναι απαράδεκτη η στάση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθυστερεί κάτι που θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει. Και μάλιστα αυτό βόλεψε πάρα πολύ, γιατί ξέρουμε ότι διαπραγματευόσασταν και τη τύπη με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Και φυσικά ενδοκρινικοί διαταράκτες εντάσσονται ε, μέσα σε αυτή τη συμφωνία καθώς οι Ηνωμένε Πολιτείε έχει μια ιδιαίτερα δευρυμένη και αποδεκτή νομοθεσία για του ενδοκρινικού διαταράκτες. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάτο. Στην κυρία Μάτο. Συγγνώμη, ε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό και αφορά την υγεία των ε, πολίτων. Προσπαθεί η Κομισιό να κάνει μια μελέτη αντικτύπου για να προσδιορίσει τα κριτήρια τα οποία αφορούν του ενδοκρινικού διαταράκτε. Ο κανονισμό για τα βιοκτώνα έθετε προθεσμία ε, στο Δεκέμβριο του 2013. Δεν απαιτεί το η μελέτη αντικτύπου από καμία νομοθεσία. Έπρεπε απλώ να σεβαστείτε τη λήξη τη προθεσμία. Η Κομισιόν που πρέπει να υπερασπίζει τι κοινοτικέ συνθήκε ακολούθησε το δικό τη δρόμο και είχαν γράψει οι βουλευτέ επιστολή στο Γιούνκερ και του υπενθύμησαν την υποχρέωση του σεβασμού των συνθήκων και ε, μάλιστα του υπενθύμησαν ότι έπρεπε η θέσπιση των κριτηρίων να γίνει το σύντομα τώρα Δεν μπορούμε να περιμένουμε τον Ιούνιο του 2016. Έτσι λοιπόν ε, σας ζητάμε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στο διάλογο με τους επιστήμονες και με το Κοινοβούλιο. Να εφαρμόσετε την αρχή της πρόληψης. Αυτό είναι προτεραιότητα πριν από οποιοδήποτε εμπορικό και οικονομικό συμφέρον. Η Κομισιόν έχει τεράστια ευθύνη απέναντι στους πολίτες που θίγονται από ε, την υπογονιμότητα και και από ενδομητρίωση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πότσακ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που ε, ε, έγιναν το 2013, Υπήρξε μια ανακοίνωση της Κομισιόν για τα επιστημονικά κριτήρια. Ε, η προθεσμία ήταν ε, ο Δεκέμβρης του 2014 και δεν έγινε τίποτα. Το 2014 η Κομισιόν δήλωσε ότι θα έκανε μελέτη επιπτώσεων. Αυτό μας δείχνει ότι η Κομισιόν στην ουσία δεν σεβάστηκε καμία προθεσμία. Ε, και ε, ούτε και τη θέση της ΕΦΣΑ. Θεωρώ λοιπόν ότι οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα πρέπει να είναι υπόλογοι εναντί των πολιτών για τις ε, πράξεις τους και να μην λένε παραμύθια. Το δικαστήριο αποφάσισε τον ε, ε, Δεκέμβρη και δεν πρέπει να συνεχίσουμε να λέμε αυτά τα παραμύθια. Ευχαριστούμε. Κύριε ε, Επίτροπε, αυτή τη στιγμή πρέπει να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι είμαι και εγώ γιατρός. 67 χρόνια ασκούσα το επάγγελμα του γιατρού. 47. 37, 37 συγγνώμη. Και πραγματικά αυτή η συζήτηση μου δείχνει ξεκάθαρα ότι ε, ε, πρέπει να είμαι ειλικρινής. Μου αρέσουν οι ειλικρινείς συζητήσεις. Και όταν λέει κάποιος ότι εγώ εκπροσωπώ τη βιομηχανία, λυπάμαι. Είναι ένα άδικο επιχείρημα. Έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές ενδοκρινολόγους, ε, τοξικολόγους, ε, βιοχημικούς. Πριν από μερικές ε, εβδομάδες συζήτησα με συμβούλους και επιστήμονες αυτό το θέμα σε μια συγκεκριμένη εξειδικευμένη συνάντηση για αυτό το θέμα. Σας προσκαλώ να έρθετε κι εσείς σε κάτι τέτοιο, γιατί πρέπει να έχουμε επιστημονικά επιχειρήματα. Ποτέ δεν θα έπαιρνα το μέρος της βιομηχανίας. Η πρώτη μου δουλειά είναι η δημόσια υγεία. Η υγεία. Και για να είμαι ειλικρινής, είμαι πραγματικά περήφανος που έχω τόσους συμμάχους εδώ που θέλουν να μαχηθούν κατά του εινοπνεύματος, ε, του, του καπνού και όλων αυτών των στοιχείων που πραγματικά βλάπτουν την υγεία των ανθρώπων. Με χαρά μου θα έβλεπα ε, αυτούς τους συμμάχους να συντάσσονται μαζί μου και σε αυτά τα ζητήματα. Είναι το θέμα αυτό δύσκολο. Πέρυσι είπαμε ότι θα γίνει μελέτη επιπτώσεων. Αυτή η μελέτη επιπτώσεων δεν έχει να κάνει με τα οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία, έχει να κάνει με τα επιστημονικά στοιχεία. Πώς ε, θα ορίσουμε τη δραστικότητα, την έκθεση, την ισχύ των ε, ουσιών αυτών. Δεν είναι εύκολο να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Πέρυσι είχαμε τρία στρογγυλές τράπεζες, είχαμε συζητήσεις, είχαμε διασκέψεις. Από πού τεκμέρεται ότι εγώ είμαι με τη βιομηχανία. Είμαι ειλικρινής, εγώ έχω πτυχίο γιατρού, είμαι υπεύθυνο, έχω ευθύνη. Ξεκινήσαμε με μεθοδολογικό τρόπο, με συζήτηση για 600 χημικά ε, υλικά που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο πραγματικά δεν ξέρω πώς να πάω πιο γρήγορα. Παρακαλώ δείξτε μου, βοηθήστε με. Είμαι κι εγώ πράσινος σαν και εσάς, όμως δεν κατηγορώ τους άλλους. Είμαι ειλικρινής και θα το πω ξεκάθαρα. Ναι, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε το συντομότερο. Αν θυμάστε πέρυσι είπαμε ότι ίσως στο τέλος του 2016 θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Τώρα σας λέω ότι θα αποφασίσουμε μέχρι το, το καλοκαίρι. Παρακαλώ, αν μπορείτε κάντε κάτι καλύτερο. Αλλά να είμαστε ανοιχτοί και διαφανείς. Και εγώ θα είμαι, αλλά να είστε κι εσείς. Σε όλα τα ζητήματα σε όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία. Να μιλήσουμε για τα ηλεκτρονικό τσιγάρο, για τον καπνό, για όλα αυτά τα πράγματα που μας περιβάλλουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά σε πολύ δύσκολη θέση όταν μιλάμε για ζητήματα δημόσιας υγείας. Είναι μεγάλο το κόστος της λιγότερης Ευρώπης στην δημόσια υγεία. Και φυσικά είμαι έτοιμος να κάνω τη δουλειά μου, αλλά πιστέψτε με, πάνω απ' όλα πρέπει Έχουμε κριτήρια τα οποία θα είναι διαχειρίσιμα, θα μπορούν να ρυθμίσουν την κατάσταση και αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι πολύπλοκο το ζήτημα. Όταν ακούω όμως τέτοια λαϊκιστικά επιχειρήματα λυπάμαι. Είμαι όμως ανοιχτός και διαφανής. Ποτέ δεν θα υποστηρίξω κάποιο λόμπι. Ποτέ δεν θα πάρω το μέρος κάποιου. Η δουλειά αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη και Πραγματικά πρέπει να συζητήσουμε με σοβαρότητα και εις βάθος πώς θα αξιολογήσουμε, πώς θα κατανοήσουμε, πώς θα προχωρήσουμε. Εγώ κάνω τη δουλειά μου πολύ καλά. Έχω χάσει ήδη ένα χρόνο και τέσσερι μήνε, όσο καιρό είμαι σε αυτή την θητεία, για να είμαι αποτελεσματικό. Αλλά είμαστε όλοι μαζί αποτελεσματικοί. Εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη δουλειά μας και να προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και να έχουμε τα κριτήρια μέχρι το καλοκαίρι. Και καλό θα είναι να ε, αποτελέσουμε και παράδειγμα γιατί είμαστε πρωτοπόροι. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη δουλειά μας βάσει επιστημονικών στοιχείων και θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε κριτήρια όσο πιο γρήγορα γίνεται ίσως το καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε για την απάντηση. Ελπίζω